Also, liebe συνάδελφοι, τώρα θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας και θα ήθελα να ε, καλωσορίσω θερμά τον Επίτροπο Τιγκέρ και σας όλους βέβαια και μπορεί να ξεκινήσει η συζήτησή μας. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω τον λόγο εις ε, τον ε, επίτροπο να μπορέσω να του δώσω το λόγο για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Αγαπητέ κύριε Ρόιλ, αγαπητοί ε, κύριοι και κυρίες ευρωβουλευτές, ε, χαίρομαι που σήμερα βρίσκομαι εδώ εις ε, την Επιτροπή για Ενεργειακά Θέματα για να παρουσιάσω την πρόσφατή μας ε, στρατηγική ενεργείας και για το πακέτο υποδομών και να έχω και τα δικά σας σχόλια και θα σας πω γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή διότι την Παρασκευή έχουμε Συμβούλιο Ενεργείας και τα θέματα αυτά θα είναι προς και εμείς ε, ούτως ή άλλως ε, ε, θα ξανασυζητήσουμε τα θέματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου για να μπορέσουμε να διαθέσουμε μισή ημέρα ακριβώς και μόνον για την ενεργειακή πολιτική κατά τρόπον ώστε η ενέργεια να συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την εξέλιξη της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης. Επ' αυτού θα βασιστούμε στο άρθρο 194 της συνθήκης της Λισαβόνας και ε, θα το παρακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Τι μας απασχολεί σε αυτή τη στρατηγική. Καταρχήν αναφερόμαστε στην εσωτερική αγορά. Η έκθεση της κυρίας Σκολάς Καμπαρίνσκα πέδειξε σαφώς όπως άλλωστε και η έκθεση Μόντι που τόνισε το συγκεκριμένο θέμα ότι έχουμε στο, στην νομοθεσία μας την εσωτερική αγορά της, του ηλεκτρικού ρεύματος εδώ και 12 χρόνια αλλά απέχουμε ακόμη πάρα πολύ από την εφαρμογή του και άρα είναι προς όφελό σα και προ συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουμε. Ποιο θα υποφεληθεί. Ε, καταρχήν ε, η Επιτροπή ε, σαν αποδέκτης αυτής της επιταγής και όντας θεματοφύλακας των συνθήκων θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Η εσωτερική αγορά είναι ύψιστη προτεραιότητά μας και έχουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις συμβατικές σχέσει με τα τρίτα κράτη και την περασμένη εβδομάδα θυμάστε ότι συμβουλεύσαμε την, ε, πολιτική, ε, την πολωνική κυβέρνηση για τα θέματα της ενεργείας προ λίγου χρόνου ε, συμβουλεύσαμε την βουλγαρική κυβέρνηση για τα θέματα αερίου και για το υπόμνημα του South Stream και άλλωστε είμαστε ουσιαστικά σε μία φάση εφαρμογής των ε, προγραμμάτων στα διάφορα κράτη και μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να προωθήσουμε ε, τα ε, ηλεκτρικά δίκτυα και θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη τα οποία ούτως ή άλλως έχουν δώσει νομική ισχύ εις τις οδηγίες και στους κανονισμούς και όλα αυτά θα συζητηθούν στις 4 Φεβρουαρίου και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν και αντιδράσεις αλλά υπάρχει μία σειρά κρατών και, ε, και κυβερνήσεων που λέγουν ότι επιθυμούν την κοινή εσωτερική αγορά, το πρεσβεύουν τις Κυριακές, αλλά όλη την εβδομάδα κάνουν το αντίθετο και αρνούνται τα πάντα. Και αυτό ισχύει για το τρίτο πακέτο της εσωτερικής αγοράς και για το ε, ανταγωνιστικό δίκαιο της Ευρώπης. Το Μάρτιο θα ξεκινήσουμε την ΕΖΑ και ελπίζω ότι ο, ο, προγραμματισμός με τη βοήθειά σας θα μπορέσει να ψηφιστεί ακόμη εντός του τρέχοντος έτους διότι χωρίς προπολογισμό δεν θα μπορούμε να αναπτύξουμε πλήρως κανένα πρόγραμμα. Η στρατηγική μας ε, μπορεί να περιγραφεί σε πέντε βασικά σημεία. Καταρχήν εξοικονόμηση ενεργείας. Για να επιτύχουμε το στόχο μας του 2020 πρέπει να μπορέσουμε να ε, υλοποιήσουμε τη δυνατότητα εξοικονόμησης της ε, ενέργειας και την αποτελεσματικότητα της ενέργειας και γι' αυτό του χρόνου το Μάρτιο θα ανακοινώσω μία νέα στρατηγική ε, για την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα και ευχαριστώ θα προσβλέπουμε στην έκθεσή σας και ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους συντάκτες εκθέσεως αυτής το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο κατά τρόπον ώστε μέχρι το Μάρτιο εμείς να διατυπώσουμε την ενεργειακή μας στρατηγική και να την υποβάλουμε και σε εσά και σε όλους τους ομολόγους μας. Δεύτερο η προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη ενεργειακών δικτύων ε, για να συνδεθούν όλα τα κράτη-μέλη και θα επανέλθω σε αυτό το σημείο και για να προωθήσουμε την, την εσωτερική αγορά. Τρίτον, ε, ασφάλεια της ε, τροφοδότησης ε, και σαφείς τιμές που μπορούν να καταβληθούν για την ενέργεια και επίσης σε ανταγωνισμό με άλλες περιοχές του κόσμου θα πρέπει να διατηρήσουμε την ε, ε, εξέχουσα θέση μας στην ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών και να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε και περαιτέρω. Και πέμπτον, όσον αφορά το γεωπολιτικό μας βάρος, θα πρέπει να ε, το χρησιμοποιήσουμε στις διαπραγματεύσεις περισσότερο, κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσουμε να ε, επηρεάσουμε περισσότερο και τους ενεργειακούς μας ομολόγους. Με τα βεβαιότητος μπορώ να πω ότι το πακέτο των ε, υποδομών είναι η βάση για την υλοποίηση των προγραμμάτων μας. Και εδώ πρέπει να εξετάσουμε το δίκτυό μας για ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο διότι έχουν παλιώσει τα δίκτυά μας και αν θέλουμε να έχουμε αλληλεγγύη, ασφάλεια και διαφοροποίηση και χρήση ε, ανανεωσίμων πληρών, πηγών ενεργείας θα πρέπει όλα αυτά να χρησιμοποιηθούν για να προωθηθεί η εσωτερική αγορά. Όσον αφορά ε, το ε, ενεργειακό πρόγραμμα για την ε, συγκυρία είναι ένα ουσιαστικό θέμα που μας απασχολεί και 97% από των πόρων θα χρησιμοποιηθούν για προγράμματα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 146 εκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για προγράμματα ανανεώσιμης ενέργειας και για ενεργειακή αποτελεσματικότητα και θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Θα χρειαστεί όμως και ενίσχυση των ε, ε, ε, των προγραμμάτων για την υποδομή στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα δίκτυα συνδέσεώς μας και να καλύψουμε όλη την Ευρώπη και θα πρέπει να πούμε επί του θέματος αυτού ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στην ε, ευρωπαϊκή υποδομή των κρατών μελών αλλά ε, υπάρχουν και άλλοι ε, συνεργάτες η Νορβηγία, η Κροατία οι υποψήφιες χώρες σαν την Σερβία και γενικώ τις χώρες των Βαλκανίων και είχαμε ήδη μία πρώτη συζήτηση ε, με τον ε, Υπουργό στο Κίεβο ε, συζητήσαμε και με την Τουρκία και η ένταξη της Τουρκίας στην ενεργειακή μας κοινότητα νομίζω θα είναι προς όφελος όλων των συμβαλωμένων μερών. Και υπάρχει μία κίνηση ε, σύμφωνα με την οποία και το Τουρκμενιστάν και το Αφγανιστάν θα συμμετάσχουν και αν ε, δούμε και την επίθεση των ε, Ρώσων ομολόγων μας βλέπουμε ότι η Ρωσία μπορεί να είναι ένας χρήσιμος συνεργάτης στα θέματα ενεργείας και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα σχέδια μαζί τους μέσα στα επόμενα χρόνια με την ανακοίνωσή μας για τις ε, ε, προτεραιότητάς μας υποδομών μέχρι το 2020 έχει ήδη γίνει ένα πρώτο βήμα. Άλλα βήματα είναι πώς θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία διοδοτήσεως, πόσο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί της διαμόρφωσης και της εφαρμογής των τιμολογίων και ε, θα συζητήσουμε όλα τα θέματα αυτά στο επόμενο έτος διότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα χρειαστούμε για τα δίκτυά μας περίπου 200 ε, δισεκατομμύρια ευρώ αλλά η ουσία είναι ε, η ιδιωτική επένδυση για να μπορέσει να πληρωθεί το κόστος της ενεργείας αλλά και κάποια συγχρηματοδότηση και αυτό θα ληφθεί η υπόψη για όλη τη δεκαετία ή στις συζητήσεις μας περί του μελλοντικού προπολογισμού. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ε, στρατηγικούς αυτοκινητοδρόμους για την ενέργεια και ε, ε, προσβλέπουμε σε μία περιφερειακή συνεργασία με ομάδες κρατών. Στην ε, βορειοδυτική Ευρώπη έχουμε τη Βόρειο Θάλασσα αλλά και στην κεντρική Ευρώπη έχουμε τα κράτη της Βαλτικής, τη Φιλανδία, τη Νορβηγία και το νοτιοανατολικό σκέλος μέχρι την Ελλάδα δημιουργούνται μεγάλες περιοχές όπου είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Στη συνέχεια θα πρέπει να βελτιώσουμε και την περιφερειακή συνεργασία με τρίτες χώρες. Και χαίρομαι διότι οι χώρες στην ε, περιοχή της ε, Βορείου Θαλάσσης ε, θα συνδεθούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των βορείων χωρών συν της Νορβηγίας μία διακήρυξη προθέσεων για να μπορέσουμε να έχουμε μία καλύτερη και πιο γρήγορη διαδικασία αδειοδοτήσεως διότι ε, όταν ε, ε, υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συντάγματα των διαφόρων κρατών να διασφαλίσουμε την νομική τάξη των εμπλεκομένων κρατών και να εξασφαλίσουμε και τα δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορούμε συγχρόνως να μείνουμε στα και να κινούμαστε πιο γρήγορα διότι η ανάπτυξη της, ε, του ανατολικού σκέλου στη δεκαετία του 90 με δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων επετράπει μόνο ε, διότι ε, μπόρεσε κανείς να κινητοποιηθεί και να ενισχύσει κατά αυτόν τον τρόπο το εμπόριο. Εάν εξετάσουμε στο διοικητικό τομέα τι τις αρχές και τα δικαστήρια βλέπουμε ότι συνήθως ε, δραστηριοποιούνται εκ των υστέρων. Δηλαδή ο ένας ζητά ε, άσυλο, ο άλλος ε, ζητά μία άδεια για οικοδόμηση και μετά έρχεται η υποδομή των, των δικτύων ενεργείας ενώ αυτά θα έπρεπε να προπορεύονται για να αποφύγουμε τη τις μακροχρόνιες αναμονές στα διάφορες, στις διάφορες φάσεις και για να μπορούμε εγκαίρως να επανδρώσουμε το σύστημά μας, να ενισχύσουμε τις τοπικές αρχές κατά τρόπον ώστε πάρα πολύ γρήγορα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αλλά συγχρόνως με απόλυτη ασφάλεια και σοβαρότητα. Χρειαζόμαστε όπως είπα ε, ένα ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο καταρχήν ε, θα επέμβει η ιδιωτική πρωτοβουλία και στο, στη συνέχεια θα μπορέσει να υπάρξει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πέραν των δύο μεγάλων αυτών πρωτοβουλειών της ενεργειακής μας στρατηγικής όπου ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργαστήκε μαζί μας πάρα πολύ ενεργά ελπίζουμε ότι το ίδιο θα συνεχιστεί και στις δύο επόμενες φάσεις και θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω την πρωτοβουλία μας ε, για τα πυρηνικά απόβλητα που θα πρέπει επίσης να συζητηθεί. Και πιστεύω ότι όσον αφορά τα πυρηνικά απόβλητα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ ψηλό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. Είναι απαραίτητη η ασφάλεια. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω και στον τομέα αυτό ήδη πριν από τις επίσημες συζητήσεις να μου μεταφέρετε τις απόψεις σας, είμαι στη διάθεσή σας για να μπορέσω να κάνω συζητήσεις μαζί σας επί του θέματος και στην Επιτροπή και ιδιωτικά διότι υπάρχουν ανάγκες βελτιώσεων και ανανεώσεων των πυρηνικών δικτύων κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα έχω μία σειρά από παρεμβαίνοντες που ζητούν το λόγο, ουσιαστικά 12 και θα έλεγα ότι επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο ίσως θα έπρεπε να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ήδη προσετέθησαν άλλοι δύο, έχουμε 14, κλείσαμε τον κατάλογο και θα σας παρακαλούσα σε ένα-δύο λεπτά να μπορέσετε να παρουσιάσετε τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Σεμάνσκι είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Δύο θέματα θα ήθελα να μας απασχολήσουν. Καταρχήν, το τι θα γίνει με την κοινή, ενέργεια, με την κοινή αγορά ενέργειας και δεύτερον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, τον ανεφοδιασμό και τη διέλευση του φυσικού αερίου μια και είναι τεράστιο ο ανταγωνισμός μεταξύ του αγωγού Ναμπούκο που είναι το ευρωπαϊκό project και του project South Stream που προωθεί η Gazprom και θα εξαρτηθεί από το ποιος θα κερδίσει αυτό το μάτς και το ποιος θα καταφέρει να χρησιμοποιήσει και θα έχει τις πιο πολλές παραγγελίες για τον αγωγό του ποια, ποιο από τα δύο μπλοκ θα είναι το πιο πετυχημένο. Πρέπει να σας πω πως αυτή τη στιγμή φαίνεται να προηγεί το South Stream γιατί προωθεί πολύ το project αυτό η Ρωσική Ομοσπονδία και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το θέμα αυτό. Υπάρχει περίπτωση να θεωρήσετε εσείς στα πλαίσια των διευρωπαϊκών δικτύων το South Stream ως project προτεραιότητας και αυτό στην εξασφάλιση του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου. Γιατί νομίζω πως αν στηρίξετε εσείς το South Stream αντί του Ναμπούκο, ο South Stream θα κερδίσει. Αναφερθήκατε σε διαβουλεύσεις που γίνονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολωνίας και της Βουλγαρίας για τους ε, αγωγούς Αμάι και South Stream. Στο Γιαμάλ, στο αέριο δηλαδή που προέρχεται από το Γιαμάλ, είναι αλήθεια πως ε, για την κοινή αγορά ενέργειας έχουμε κάποιους περιορισμούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κύριε Επίτροπε και για την παρουσία σας εδώ και για την ε, περιοκτική σας εισήγηση. Συμφωνούμε μαζί σας ότι το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ενέργεια στις 4 ε, Φεβρουαρίου δίνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για την υψηλή προτεραιότητα που έχει πλέον η ενέργεια, η ενεργειακή πολιτική στη βάση του άνθρου 194 της Συνθήκης. Ελπίζουμε πραγματικά ότι και τα αποτελέσματα αυτού του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα δικαιώσουν ε, αυτήν την, ε, την επιλογή και αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως ελπίζουμε και βασιζόμαστε σε εσά ότι θα διατηρήσετε διαρκή και ισχυρή την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικά αυτής της Επιτροπής σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και διεξαγωγής των συζητήσεων για αυτό το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Επίτροπε. Στην ε, νέα ενεργειακή στρατηγική για το 2020, ε, η Επιτροπή θέτει ως στόχο την εξασφάλιση ενός απαραίτητου βαθμού σύγκλησης ή εναρμόνισης των εθνικών καθεστώτων στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποστηρίζοντας, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η αγορά μετατρέπεται από τοπική σε, σε διασυνοριακή. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι τα κράτη-μέλη και, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα έχουν υποστηρίξει με θέρμη το ισχύον καθεστώς ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των ανεξάρτητων εθνικών καθεστώτων στήριξης και με, από μια πρώτη ανάλυση των ε, εθνικών σχεδίων δράσης που έχουν υποβληθεί προκύπτει ότι πήραμε τη σωστή απόφαση νομίζω καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τεσσάρων χωρών αν θυμάμαι καλά, ε, δηλώνουν ρητός και αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να καλύψουν τους ε, στόχους τους για το 2020 από εγχώριες πηγές. Ανησυχούμε λοιπόν μήπως μία πρόορη προσπάθεια αλλαγής αυτού του πετυχημένου μοντέλου τα επόμενα χρόνια ε, με τη δημιουργία αγοράς πράσινων πιστοποιητικών θέσει σε κίνδυνο την ισόρροπη ανάπτυξη αποκεντρωμένων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. και ε, επίση, και τελειώνω κύριε Επίτροπε, αναγνωρίζετε κι εσεί και μέσω τη ανακοίνωσή σα, ότι ένα μοντέλο διασυνοριακή προώθηση των ΑΠΕ προϋποθέτει και τι κατάλληλε ενεργειακέ υποδομέ, για τι οποίε απαιτούνται μεγάλε επενδύσει σε βάθο χρόνου. Υπογραμμίζεται αυτό στην ανακοίνωσή σα για το πακέτο των υποδομών. Θέλω λοιπόν να σα ρωτήσω πώ σκοπεύετε να ε, αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα και αν σκοπεύετε να αναθεωρήσετε την οδηγία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα στα επόμενα χρόνια, ώστε ε, να προχωρήσετε αυτή την ιδέα της εναρμόνισης των εθνικών καθεστώτων στήριξης μέσω της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας πράσινων πιστοποιητικών. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, είπε η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς κύριε Επίτροπε για μια τόσο σφαιρική παρουσίαση. Με χαρά αναμένουμε τη στενή συνεργασία που θα έχουμε μαζί σας τους επόμενους μήνες. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ασχολήθηκα με το θέμα της αποδοτικότητας σε ενέργεια και θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για το πακέτο των ευρωπαϊκών υποδομών. Είναι ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας, το είπατε κι εσεί, και ξέρετε πω η δική μου ομάδα θεωρεί πω η ανανεώσιμη ενέργεια είναι μία από τι προτεραιότητε οι οποίε θα πρέπει να προωθήσουμε και στα πλαίσια τη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για να εξασφαλίσουμε τον ενεργειακό ανεφοδιασμό των κρατών μα. Ξέρω πω αρκετά κράτη-μέλη έχουν μετακινηθεί προ άλλοι είδε πρωτοβουλίε, αλλά όλοι στι ανανεώσιμε έχουν πολλά project στα σκαριά και θα ήθελα να δούμε αν υπάρχουν ευρωπαϊκέ υποδομέ που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στι προκλήσει τη ανανεώσιμη ενέργεια. Καταρχήν έχουμε αυτό το σούπερ δίκτυο το ηλεκτρική ενέργεια το οποίο αναφερθήκατε, το οποίο εξασφαλίζει πω μεγάλα σχέδια ε, ανανεώσιμη ενέργεια θα μπορούσαν να τροφοδοτούν το ηλεκτρικό μας δίκτυο. Έτσι θα έχουμε λοιπόν μαζική τροφοδοσία. Και το άλλο είναι η ευφυής τα ευφυή δίκτυα, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε προ... ενέργεια που πρέπει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούμε άμεσα να την τροφοδοτήσουμε στο δίκτυό μας. Αυτό που μου έχουν καταγγείλει είναι ότι πολύ Πολλές φορές οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την πρόσβαση στην αγορά. Ε, τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στο δικό μου κράτος. Ποιε πρωτοβουλίες λοιπόν μπορείτε να λάβετε έτσι ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργεια από ανανεώσιμε πηγές να μπορούν εύκολα να τροφοδοτήσουν το δίκτυο. Έτσι ώστε αυτό το είδο τα FEE δίκτυα ε, να τροφοδοτούνται ε, χωρίς δυσκολίες κυρία Χέρτσοκ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση, η οποία ήταν πάρα πολύ πληροφοριακή και νομίζω ότι καλό θα ήταν να έρχεστε πιο συχνά να μας βλέπετε, να είστε σίγουροι πως εμείς στις προσπάθειές σας σας στηρίζουμε. Καταρχήν για την 4η Φεβρουαρίου που θα γίνει μια διάσκεψη υπό Ουγγρική Προεδρία, πείτε μου ποια είναι τα ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτή τη σύνοδο. Και πώς θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας βοηθήσει για να εξασφαλίσετε την επιτυχία αυτής της συνόδου. Δεύτερον, τι περιμένετε για να υποβάλλετε προτάσεις για τις ευρωπαϊκές υποδομές. Για τεφή αυτά δίκτυα τα οποία θα έχουν τη μέγιστη δυνατόν αποδοτικότητα. Νομίζω πως θα πρέπει εδώ να προσέξετε γιατί τα δίκτυα αυτά θα έρθουν σε, άμεση, σε άμεσο ανταγωνισμό ε, με ε, τις κλασικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές τους. Και τρίτον, μια παρατήρηση περισσότερο και όχι ερώτηση. Χαίρομαι που είχατε το θάρρος να υποβάλλετε αυτή την πρόταση για τις ανανεώσιμες πηγές και σας ε, εξασφαλίζω πως οι συζητήσεις που θα γίνουν εδώ στο Κοινοβούλιο θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire. Ευχαριστώ πολύ, λέει κύριο Σενά, για τη μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημιουργία ε, μιας ευρωπαϊκής ε, ε, αγοράς ενέργειας. νομίζω ότι θα φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε καλές τιμές και αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Ο νόμος αυτός ε, που το λένε όλοι φωτισμένοι και έξυπνοι εμπειρογνώμονες θα καλύψει το μερίδιο 7 με 11% της αγοράς και μέχρι το 2015 θα φτάσει αυτό στο 21%. Οι εμπειρογνώμονες λένε πως θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη πως υπάρχει ο κίνδυνος και το υπογραμμίζουν οι εμπειρογνώμονες να είναι οι ενδιάμεσες εταιρείε οι οποίες θα έχουν τα μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη σε αυτή την περίπτωση. Σας ρωτώ λοιπόν τι μέτρα θα πάρετε για να αποφύγει το καταναλωτής ε, να πέσει θύμα αυτών των μεσαζόντων. Αυτό που πρέπει να προωθήσουμε είναι το γενικό συμφέρον για να εξασφαλίσουμε τον αναφοδιασμό όλων, να μην έχουμε στήρο ε, και αποτρεπτικό ανταγωνισμό. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκρίνουμε το κόστος έτσι ώστε να επιμεριστεί, ε, να επιμεριστεί το κόστος επένδυσης στην ανάπτυξη και ε, να εξασφαλίσουμε καλές τιμές στον καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, λέει ο κύριος Μπαλτσίτης, κύριε Επίτροπε, για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που ήρθατε, αλλά να σας ευχαριστήσω και για την ανακοίνωση αυτή που μας διαβάσετε, η οποία πιστεύω πως ήταν εξαιρετικά σαφής. Νομίζω ότι αν την είχατε παρουσιάσει πριν από ένα χρόνο, ενδεχομένως να μην την είχαμε καταλάβει κιόλας, αλλά η κατάσταση μεταλλάσσεται και πρέπει να κάνουμε κάποιες προβλέψεις για το μέλλον, όπου πιστεύω πως θα έχουμε ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο ενεργειακό σύστημα έχει το σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει ένα νέο ενεργειακό χάρτη για την Ευρώπη και νομίζω πως σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα εθνικά ενεργειακά σχέδια και πώς αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. Κάποια κράτη αντιμετωπίζουν το εξή δίλημα. Να ξεκινήσουν με την κατασκευή και οικοδόμηση μεγάλων εγκαταστάσεων, για παράδειγμα τύπου πυρηνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή όχι. Η απάντηση δεν είναι πάντα τόσο σαφής όσο θα θέλαμε και ίσως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει ε, κάποιες συμβουλές στα κράτη-μέλη για τις επιλογές που θα κάνουν. Έχουμε πει πως πολλές φορές είναι φθηνότερη η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται πυρηνικά από αυτή που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θα συμφωνήσω όμως και εσείς μαζί μου πως είναι απαραίτητο να δώσουμε κάποια κίνητρα στα κράτη που θα χρησιμοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές περισσότερο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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα κύριε Επίτροπη να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις ιδίω πριν από το Συμβούλιο Ενεργείας. Για μένα είναι πολύ βασικό να αναπτύξουμε την ενεργειακή υποδομή, άλλωστε το αναφέρατε κι εσείς και είμαι επιφυλακτική όσον αφορά τη χρηματοδότηση γιατί είπατε ότι ένα μέρος θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά, ένα μέρος θα συγχρηματοδοτηθεί αλλά έχουμε την συζήτηση του προπολογισμού και τις συζητήσεις για τον προπολογισμό στα κράτη-μέλη και αντιλαμβάνουμε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα και θα πρέπει ίσως το θέμα αυτό να θυγεί για να δούμε πόσο θα χρηματοδοτηθούν καλύτερα τα ενεργειακά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη διαδικασία της αδειοδότησης θεωρώ ότι είναι πήγον και σας ευχαριστώ ότι προχωράτε τόσο αποφασιστικά διότι το θέμα της αδειοδοτήσεως είναι ε, κάτι το οποίο πηγαίνει ομαλά. Βέβαια στην ε, Γερμανία έχουμε κάποια προβλήματα. Πώς μπορούμε να επέμβουμε ε, χωρίς όλοι να επικαλεστούν την επικουρικότητα και ότι είναι κάτι το οποίο δεν σας απασχολεί και μπορεί να ρυθμιστεί εκτός Ευρώπης. Επίσης για το 4T ήθελα να ρωτήσω εάν θα συμμετάσχει στα ενεργειακά προγράμματα, αν είναι μία προτεραιότητα και τι συγκεκριμένο σκέφτεστε να κάνετε για να προωθήσετε αυτό το τόσο σημαντικό ενεργειακό πρόγραμμα. Ο Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο γιατί θα επαναλάβω την ερώτηση Αγγέλικα για τη χρηματοδότηση. Κύριε Επίτροπε, που κατά τη γνώμη μας είναι ζωτική για να εξασφαλίσουμε αυτά τα οποία εσείς μας παρουσιάσατε. Όταν λοιπόν αναφέρεστε σε νέο χρηματοδοτικό μέσο, νομίζω πως αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτά τα ευρωομόλογα και να είναι αυτά τα εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Έχετε όμως κάποιο χρονοδιάγραμμα στο μυαλό σας για το πότε αυτό το μέσο θα εμφανιστεί, τι θα είναι, ε, θα είναι ευρωομόλογα, θα είναι κάποια εγγυημένα δάνεια για τις δημόσιες αρχές, πώς ακριβώς θα γίνει και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να σας ε, θα ήθελα να συζητήσουμε είναι η διαδικασία διοδότησης, γιατί και αυτή πρέπει να είναι σαφής. Μιλάτε λοιπόν για αυτή την ενιαία θηρίδα στην οποία απευθύνεται κανείς μόνο και μόνο για να μπορεί να λύσει σε ένα σημείο όλα τα θέματα σχετικά με τις άδειε και το συντονισμό μεταξύ περιφερειακών, κρατικών και τοπικών αρχών. Είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και θα το στηρίξουμε ε, όταν το προτείνετε γιατί αυτή η μέθοδος νομίζω είναι η μόνη που θα εξασφαλίσει όλα αυτά τα σχέδια υποδομών. Αυτές όμως λοιπόν τις θηρίδες ε, άμεση εξυπηρέτηση πώς θα τις ε, δρομολογήσετε και πώς θα εξασφαλίσετε ότι η διαδικασία αυτή θα κλείσει μέσα σε μια πενταετία και από πότε ξεκινάει να τρέχει η πενταετία, από το 2014, το 2018, τι θεωρείτε εσείς μια ρεαλιστική ημερομηνία έναρξης. Κύριο Στούρμες, διαδικαστικό. Νομίζω ότι μετά από αυτές τις ερωτήσεις που έχουν ήδη τεθεί καλό θα ήταν να μπορέσει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να, να ερωτηθούν ε, τα επόμενα θέματα διότι δεν είναι δυνατόν και δεν θα υπάρχει ίδια δυναμική. Ε, ήθελα να δώσω σε όλους τους συναδέλφους τη δυνατότητα να επέμβουν αλλά δεν έχω πρόβλημα εάν θέλετε να σταματήσουμε τις ερωτήσεις τώρα θα μπορέσει ο ο, ο, Επίτροπος να δώσει μία πρώτη απάντηση και μετά θα μιλήσει ο κύριος Ζαντό. Τώρα είναι δικό σας πρόβλημα. Εσείς τι έχετε να πείτε. Κάθεστε δίπλα στον κύριο Τούρμες. Όσον αφορά τους αγωγούς του αερίου και τον, ε, ε, την διέλευση δεν θέλουμε να μπλοκάρουμε ούτε να καθυστερήσουμε το πρόγραμμα South Stream. Εμείς θεωρούμε ότι το South είναι ένας αγωγός ο οποίος καταρχήν θα πρέπει να μεταφέρει ε, αέριο από την ε, Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να το διαφοροποιεί. Οι δυνατότητες ε, του αερίου που θα έρχεται από τη Ρωσία έτσι θα βελτιωθούν. Δεν είναι δηλαδή ένας αγωγός ο οποίος θα επηρεάσει το περιβάλλον στο χώρο από τον οποίο θα κινηθεί. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι το TAP και το ITGI νότια είναι τα μικρότερα προγράμματα και πρέπει να πιέσουμε συγχρόνως και το μεγαλύτερο το Ναμπούκο στην κεντρική Ευρώπη. Ε, όσον αφορά το θέμα του Αζερβαϊτζάν ε, δεν υπάρχει αλλαγή, είναι έτοιμο να μας προσμηθεύσει. Ε, υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί η δυνατότητα της Αυστρίας μέσω των χωρών μέσω Βουλγαρίας και μετά προς Ανατολάς είναι δεδομένη ε, το θέμα προς συζήτηση είναι ο όγκος της προμήθειας και πιστεύω ότι θα πρέπει καταρχήν στη Βαγδάτη να υπάρξει μία κυβέρνηση η οποία να δραστηριοποιηθεί και να μπορέσει να αποτελέσει μία βάση με την οποία να συζητήσουμε και επίσης ο πρόεδρος του Τουρκμενιστάν πρόσφατα διεκήρυξε την θέλησή του να μας προμηθεύσει και να δημιουργήσει μία, ε, ε, έναν αγωγό ο οποίος θα είναι υποθαλάσσιος και θα φτάσει σε μας. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, υπάρχουν τεκμηριωμένα αυτά τα ε, και οι δηλώσεις και ίσως διαβάσατε ότι ο κύριος Πούτιν, ε, ο αρχηγός της κυβερνήσεως της Ρωσίας ήταν στο Βερολίνο, έκανε ενδιαφέρουσες προτάσεις για την βιομηχανία και το εμπόριο αλλά πολύ επιφυλεκτικός για το, την ενεργειακή εσωτερική αγορά ότι έχουμε τις σχέσεις Πολωνίας-Ρωσίας, Βουλγαρίας-Ρωσίας και βλέπουμε ότι ε, η ρωσική κυβέρνηση διεξήγαγε προ λίγων ημερών τον δέκατο διάλογο με την Ευρώπη ε, και πρέπει να διευκρινίσουμε τη φιλοσοφία μας ή στους Ρώσους ομολόγους μας ε, να εξασφαλίσουμε ότι θα καλυφθούν και τα δικά του συμφέροντα. Ο κύριος Πούτιν δεν είναι πολύ θετικός. Ε, είπε ότι αν κάνετε αγωγούς θα τους τρυπήσουμε. Ε, δεν ήταν πολύ λογικός, ήταν πιο πολύ έτσι εύθυκτος και συγκινησιακός, συγκινησιακά οθούμενος. Ε, εάν συμφωνήσετε πριν από την 4η ε, ε, Φεβρουαρίου θα επανέλθω στην Επιτροπή σας κατά τρόπον ώστε να παρουσιάσω και να συζητήσω μαζί σας την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Θα έχουμε μία συνάντηση με τον πρόεδρο Φων και όταν ε, θα υπάρχουν όλα τα έγγραφα θα προσαρμοστούμε εις τις υποδείξεις του κυρίου Ρομπόη και Μπαρόζο. Καταρχήν πρέπει να γίνει μη ένας ενδιάμεσος απολογισμός, να θίξουμε τα θέματα της ενεργειακής υποδομής, να διατυπώσουμε μια ενεργειακή πολιτική προς τα τρίτα κράτη, δηλαδή μια ενεργειακή εξωτερική πολιτική, ενεργειακή έρευνα και ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι τα πέντε θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε 10 χρόνια εκεί που προσβλέπουμε. Το θέμα που άπτεται της εναρμόνισης των κανόνων για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας εφόσον έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς την προηγούμενη δεκαετία σε πάρα πολλά ε, κράτη ε, κανόνες και ε, συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν να αναπτυχθούν οι πηγές ανανεώσιμων πηγών ενεργείας πρέπει τώρα να επεκταθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρομαι στο το αιωλικό πρόγραμμα εις τη βόρεια, στις βόρειες ακτές της, του Ηνωμένου Βασιλείου, στην Ορβηγία ε, εις ε, τα προγράμματά μας για Μητροπόλεις όπως ε, το Αμβούργο, το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και όλα αυτά θα υπερβούν την, τον χώρο κυριαρχίας ενός κράτους μέλους οπότε θα πρέπει για τις αποθηκεύσεις και για τις τιμές να συζητήσουμε διασυνοριακά και αυτό είναι πολύ πιο σαφές για τις ρυθμίσεις στη Μαύρη Θάλασσα στην ε, Βόρειο Θάλασσα. Οπότε ε, μία εναρμόνιση των κανόνων για τις προτεραιότητες και για την τιμολογιακή πολιτική είναι πολύ σημαντική διότι ε, η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί με ένα διαβατήριο ή με ένα έγγραφο. Πρέπει λοιπόν να γίνουν ρυθμίσεις μακροπρόθεσμες για τα διασυνοριακά ευρωπαϊκά προγράμματα και αυτά δεν υπάρχουν επαρκώς ακόμη. Έχουμε δημιουργήσει μία task force η οποία το αργότερο την άνοιξη θα απαντήσει στο ερώτημα του τι πρέπει να κάνουμε σαν Ευρωπαίοι. Και νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να τυποποιήσουμε την τεχνική, δηλαδή να δούμε ε, τι όψη πρέπει να έχουν ε, οι Επίση, ε, Επίσης πρέπει να δούμε ε, πώς η ε, ΕΚΤ και η ICT θα μπορέσουν να συνεργαστούν. Έχουμε το θέμα Smart Cities και το θέμα των δικτύων για ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και προστιθέμενη αξία. Έχουν γίνει ενδιαφέρουσες προτάσεις επ' αυτών των θεμάτων και ελπίζω ότι ιδίω όσον αφορά το πρόγραμμα Φάρος που είναι το Smart Cities θα μας στηρίξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα της εσωτερικής αγοράς πιέζουμε και όταν τελειώσουν οι προθεσμίες για το τρίτο πακέτο του χρόνου θα πρέπει ε, να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για τα διαδοχικά προγράμματα ε, διότι ορισμένες γενικές ε, διευθύνσεις τώρα συζητούν με τα κράτη-μέλη όπου χρειάζονται οι αναγκαίες νομοθετικές ε, διατυπώσεις. Αναφερθήκαμε, αναφερθήκατε στη χρηματοδότηση και την αδειοδότηση. Για τη χρηματοδότηση καταρχήν θα πρέπει η, ε, ε, τα εθνικά ρυθμιστικά νομοθετήματα για τη διαμόρφωση των, τιμών να διεκπαιρεωθούν εθνικά. Αυτό είναι το πρώτο έργο για να μπορέσουν να προωθήσουν τον ανταγωνισμό, να αποφύγουν τα καρτέλ και δεύτερον να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα μέσα στο οποίο θα υπάρχει σταθερότητα των τιμών. Υπάρχει βέβαια εδώ και ένα στοιχείο αύξησης των τιμών διότι υπάρχει η τιμή για τους ιδιοκτήτες, ε, υπάρχει αδειοδότηση, ε, υπάρχει επίσης η προσθήκη ε, για κάποιο απόθεμα με το οποίο να μπορέσει να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί ή να ανανεωθεί το δίκτυο και παρόλα αυτά το σύστημα που είναι αρκετά περίπλοκο θα πρέπει να βρει ευρωπαϊκές λύσεις και σύγχρηματοδότηση για να αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι αυτά μου τα σχόλια είναι προσωπικά και όχι ακόμη επίσημα. Όταν το πρόγραμμα συγκυρίας το οποίο έχετε διατυπώσει για τρία χρόνια και αποβλέπει στην ενεργειακή υποδομή και θα χρηματοδοτηθεί με 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα αποτελέσει μια καλή βάση και με ποσοστά συγχρηματοδοτή από 10 έως 40% ιδίω στο διασυνοριακό τομέα και για τις μικρότερες χώρες όπου οι αγορές και οι χρήστες δεν είναι ακόμη τόσο ισχυροί. Δηλαδή θα υπάρχουν 800 εκατομμύρια ε, το χρόνο και αυτά θα ε, ενσωματωθούν στην επόμενη ε, περίοδο και θεωρούμε ότι είναι λογικό να υπάρξουν για την επόμενη οχταετία, δεκαετία για τις χρηματοδότηση της υποδομής, όχι μόνο την εποχή της κρίσεως αλλά και σε, φυσιολογικά, σε φυσιολογικές οικονομικές κρίσεις. Επίσης ε, όσον αφορά τον ε, προγραμματισμό προσβλέπουμε εις ε, τους συνεργάτες μας και ομολόγους οργανισμούς και ε, θα πρέπει να υπάρξει μία ε, επιτάχυνση των ε, διαδικασιών, των προγραμματισμών για την νομοθετική προώθηση, για την αδειοδότηση, για την τιμολογιακή πολιτική, αλλά όλα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν μόνο σε εθνικό επίπεδο. Και θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην προώθηση της ενεργειακής δις υποδομής ε, να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές κατά τρόπον ώστε ε, τα εθνικά κράτη ε, να κρατήσουν την κυριαρχία τους και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να μπορέσουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να προωθηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε διαχερσαία οδού αντί σε 20 χρόνια σε 8 ή 10 χρόνια. Όλα αυτά είναι θέματα που απασχολούν την ενεργειακή πολιτική. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω και για το χώρο της Μεσογείου γιατί οι Γάλλοι τώρα έχουν δημιουργήσει μία ομάδα και πρέπει να δούμε εάν με Ευρωπαίους επενδυτές μπορούμε να συνεργαστούμε ή στη Λιβύη, στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τινησία και αργότερα και με άλλες χώρες. Εάν μπορούμε να προκαλέσουμε εκεί επενδύσεις κατά κατά τρόπον ώστε να χρησιμοποιήσουμε ε, το ρεύμα και σε αυτές τις χώρες υποδομή για την ηλιακή ενέργεια, για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τη θέρμανση, την ψήξη, να χρησιμοποιήσουμε ε, το νερό της θάλασσας, την ε, υδραυλική ενέργεια και να εναρμονίσουμε μία ακόμη φορά το Ευρωπα... την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία νομοθεσία και ε, την νομοθεσία των κρατών μελών στον τομέα των ε, ανανεωσίμων ενεργειών. Δηλαδή ε, η ισπανική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και η ανάλογη γαλλική να γίνουν μια ευρωπαϊκή που θα συνδέεται μέσω των πυρηναίων διότι αυτό το πρόγραμμα δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Τώρα ο κύριος Ζαντό έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Αναφέρατε ως ε, προτεραιότητα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και μετά μπήκαμε στη συζήτηση για τους αγωγούς και την προμήθεια σε φυσικό αέριο. Να υπενθυμίσω ότι το 20% της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη είναι το ισοδύναμο με 15 αγωγούς Ναμπούκο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Επίσης αναφέρατε το πρόγραμμα επισκέψεων του Προέδρου Μπαρόζο ε, στην ε, περιοχή, ε, στις περιοχές που θα μπορούσαν να μας προσφέρουν φυσικό αέριο, θεμητό είναι. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το Φεβρουάριο στη Σύνοδο Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στον τόπο που θα γίνει αυτή η σύνοδο, θα είναι θα γίνει μία έκθεση ε, με, τα, με, τις καλύ, τους καλύτερους καυστήρες που μπορούμε να έχουμε στην ευρωπαϊκή αγορά, πέρα από τις ομιλίες δηλαδή. Ε, γιατί αν μπορούσαμε μέσω της, ε, του design να βελτιώσουμε την επίδοση, την ενεργειακή, τις των καυστήρων, ε, θα φτάσαμε στο 10% της μείωση. θα μειώναμε την κατανάλωσή μας ενέργεια κατά 10%. Μιλήσατε για την, μιλήσατε για την ενεργειακή φτώχεια. Πολύ σημαντικό θέμα. Δεν περιορίζεται μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια. Αν είχαμε ε, στο θέμα των νομοθετημάτων ε, που υπάρχουν για το διοξείδιο του άνθρακα, για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, αν, είχαμε, αν ήμασταν φιλόδοξοι, θα μπορούσαμε να μειώσουμε κατά 20-30% την κατανάλωση καυσίμων από τα αυτοκίνητα. Το ίδιο αν είχαμε μια, μια πραγματική πρωτοβουλία για τα κτίρια, με την ανακαίνιση των υπαρχών των κτίριων. Θα μπορούσαμε δηλαδή σε πολλά κτίρια να μειώσουμε κατά 2 ή κατά 3 το λογαριασμό του ηλεκτρισμού. Δεν, μπορούμε, δεν πρέπει δεν, να, κάνουμε, να καταστήσουμε προτεραιότητα την επένδυση σε αυτού του τομεί. γιατί ναι μεν καλοί είμαστε στα λόγια ω προ φιλοδοξίες, αλλά δεν περνάμε ποτέ στα έργα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μετσάρος. Η ενεργειακή πολιτική είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σας ευχαριστούμε βεβαίως πραγματικά θερμά, Επίτροπε, για τις ε, ευθύνες σας και για την προσπάθεια εναρμόνισης, όπου κάνετε ό,τι μπορείτε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο ενεργειακός ανεφοδιασμός είναι πολύ σημαντικός και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη σχετική έκθεση. Ε, είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που σήμερα εξαρτώνται πάρα πολύ από αλλού και είναι και πολύ ευάλωτες σε αυτόν τον τομέα της ενέργειας. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ε, επίτροπε, σύν το χρόνο θα καταφέρουμε να εντάξουμε στις ευρωπαϊκές ε, υποδομές τις χώρες που μπήκαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004. Θα τις εντάξουμε λοιπόν αυτές τις χώρες. Μιλάμε τώρα δηλαδή για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το θέμα είναι οικονομικό, αλλά έχετε μια ιδέα για το χρονοδιάγραμμα ένταξης αυτών των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Χαίρομαι που εσχάτως ε, καταφέραμε να μιλήσουμε πιο ειλικρινά για, την για τα πυρηνικά. Νομίζουμε ότι θα μπορούσαμε να εφοδιαστούμε από πυρηνικά εργοστάσια με ενέργεια κατά 40 με 45%. Ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλά επίτροπες σε αυτό το τομέα. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά με κάθε ασφάλεια των πυρηνικών αποβλήτων. Ποια είναι η γνώμη σας, Πρόεδρε. Επίσης θα πρέπει να ζητήσουμε την ε, συνένεση των κοινοτήτων από τις οποίες διέρχονται αυτά τα καύσιμα, ούτω ώστε να μην ε, επαναληφθούν αυτά που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα κατά τη μεταφορά επικίνδυνων ε, πυρηνικών αποβλήτων. Επίσης, τι γνώμη έχετε για την έρευνα και ανάπτυξη. πού θα δίνετε τα περισσότερα χρήματα, σε ποιο τομέα ακριβώ. Μία. Ούντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για τη σημασία που δίνετε στην Επιτροπή μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι και κοινοτικοποίησαμε την οργάνωση της αγοράς και το θέμα της ασφάλειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ένα ερώτημα για την αγορά ενέργειας. Η οργάνωση της αγοράς αυτής ενέργειας. Δεν μπορούμε ε, να έχουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά δεν υπάρχουν ρυθμιστικέ ευρωπαϊκέ αρχέ. Μιλήσατε, για, έχουμε μιλήσει μάλλον για ρυθμιστικέ αρχέ στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Πώ μπορούν οι, εθνικοί, οι εθνικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές, ρυθμιστικές πάντα, να συνεργαστούν. Επίσης, στην ε, περιοχή της Κασπίας ε, υπάρχει αυτό το εργοστάσιο φυσικού αερίου. Ήταν μια παλιά ιδέα. Σήμερα που βρισκόμαστε, η οποία μοιάζει να μην ευθυγραμμίζεται πολύ με, την, με τους ανταγωνιστικούς προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ερώτηση για την Desertec. Πού έχει φτάσει αυτό το θέμα, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Και τελευταίο θέμα για τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Εποπτεύεται ποιος είναι ιδιοκτήτης. Εμείς οι πολίτες μπορούμε να έχουμε τη διαβεβαίωση καθώς θα απελευθερώνουμε την εσωτερική μας, τον τρόπο που λειτουργεί η εσωτερική αγορά ενέργειας, ότι κανένας ξένος operator δεν μπορεί να γίνει διοκτήτης ενός τμήματος δικτύου φυσικής ενέργειας ή α, ηλεκτρισμού. Φαντάζομαι, ας πούμε, μιλάω τώρα για, για κάποιο Κινέζο, ας πούμε, για την Gazprom, να έρθουν εδώ πέρα και να μας αγοράσουν, ας πούμε. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Ε, Τούρμες. Καταρχήν ε, θα ήθελα να αναφερθώ στα σχόλια της κυρίας ε, Νίμπλερ σχετικά με την ε, υποδομή την οποία θα πρέπει να συνδυάσουμε. Έχω μία ερώτηση στην οποία θέλω να θίξω. Την ε, δήλωση την οποία κάνατε για την εναρμόνιση των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας και να σας υπενθυμίσω ότι το φθινόπωρο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει ένα πρότυπο ε, για μία εναρμόνιση σε όλη την Ευρώπη βάσει πρασίνων πιστοποιητικών. Σαν ε, βουλευτές τότε τότε το είχαμε αναλύσει και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καταρχώς, ε, ε, καταρχήν αν έχουμε ε, εθνικά δεσμευτικά συστήματα θα, θέλαμε, θα ήθελαν τα κράτη να ρυθμίσουν το θέμα εθνικά. Η Πολωνία ποτέ δεν είχε δεχτεί αυτή την οδηγία διότι δεν ήθελε να αναπτυχθεί κάτι στο έδαφος της, να αφαιρεθεί μετά και να χρειαστεί να επενδύσει η Πολωνία εκεί. Μετά, όταν μιλάμε για εθνικά συστήματα fit-in ή συστήματα με συγκεκριμένα πιστοποιητικά, θα δημιουργήσουμε μία αγορά οριακού κόστους και για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την νεολική ενέργεια θα έπρεπε να πληρώσουμε τα πάντα και θα ήταν πολύ πιο ακριβό κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια για τους πολίτες. Έτσι όμως που ε, εσείς το εξηγήσατε φοβάμαι ότι ξανανοίγεται μια συζήτηση στην οποία έχουμε κάνει πολύ, πολύ ε, ουσιαστικά ότι επιτίθεστε στα εθνικά συστήματα και ε, την για στην οδηγία, στον κανονισμό για ε, ε, τι ανανεώσιμε ανανεώσιμες πηγές ενεργείας που δεν ισχύει ακόμη, θα ισχύσει από 5 Δεκεμβρίου. Πρέπει λοιπόν να μου πείτε τι γίνεται, διότι έχουμε διάφορους μηχανισμούς ή στον κανονισμό αυτό που λέγεται ότι μπορούμε ε, με την offshore wind μπορούμε να κάνουμε τα εξής μέσω του κανονισμού και για τα 300 ή 500 ΜΒ τα οποία ουσιαστικά μιλάμε που ουσιαστικά είναι πενταροδεκάρες σε αυτό το, σε αυτό το θέμα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε και δεν ε, πρέπει ε, να διακινδυνεύσουμε ε, τα εθνικά προγράμματα για ένα πρόγραμμα 300 ΜΒ. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι που παίζετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η κυρία μέρκη είναι η επόμενη. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Μιλήσατε προηγουμένως για τους ευφυείς μετρητές. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για, τους, ε, για την ε, τοπική παραγωγή ενέργειας. Μιλήσαμε επίσης και για τις ευφυείς πόλεις. Και το άλλο είναι τα πρότυπα. Με σοκάρει το γεγονός πως τα πρότυπα εμφανίστηκαν τόσο αργά στο λόγο της Κομισιόν. Μιλήσαμε για ηλεκτρικά οχήματα, τα ηλεκτρικά οχήματα τα συζητάμε από την αρχή της χρονιάς, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει τώρα πως θα παρουσιάσει πρότυπα το 2012. Τι είδους πρότυπα είναι αυτά τα οποία περιγράφεται και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη τα οποία ε, θέλουν να έχουν αυτούς τους ευφυείς μετρητές και στο παρελθόν για λόγους προστασίας του ιδιωτικού χώρου ε, η δική μου χώρα ήταν κατά. Επίσης μιλήσαμε για το σούπερ δίκτυο. Εγώ δεν έχω δει κανένα σχέδιο το οποίο να παρουσιάζει μια σφαιρική προσέγγιση στο θέμα αυτό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πως η τοπική παραγωγή ενέργειας θα είναι διαθέσιμη μέσω interconnections. Εμείς μιλάμε για σούπερ αυτοκινητοδρόμους, εντάξει. Ίσως όμως αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι σούπερ ε, αυτοκινητόδρομοι για την ηλεκτρική ενέργεια. Μια και επαναλαμβάνω έχουμε και την τοπική παραγωγή σε μικρότερο όγκο. Καλό είναι λοιπόν να προωθήσουμε την τοπική παραγωγή και την μικροπαραγωγή ενέργειας. Ξέρω πως ε, ήταν πολικές οι θερμοκρασίες σήμερα στις Βρυξέλλες και νομίζω ότι μπορεί να είδατε και πιγκουίνους να καταφθάνουν στις πόρτες της Κομισιόν, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν μια διαφήμιση για τον ε, φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό γιατί είπαμε μέχρι το 2020 40 δισεκατομμύρια μπορούν να εξοικονομηθούν αν βελτιώσουμε τα θερμοσύφωνα και τους λέβητες. Άρα λοιπόν αυτή η αποδοτικότητα ενεργειακή είναι ένας καταπληκτικό τρόπος όχι μόνο να μειωθεί το κόστος για τον καταναλωτή αλλά για να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός για να επιτύχουμε τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή. Πότε λοιπόν θα γίνει δεσμευτική αυτή η υποχρέωση για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ε, Κύριος Γκίρεκ, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Νομίζω πως οι θερμοκρασία στις Βρυξέλλες και ο καιρός στις Βρυξέλλες είναι το αποτέλεσμα όχι μόνο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και κάποιων άλλων παραγόντων. Έχω τώρα τρεις ε, ερωτήσεις που θα ήθελα να απευθύνω στον Επίτροπο. Το 3 επί 20. Αυτό είναι ένα στόχο τον οποίο καλό θα ήταν να επιδιώξουμε με ευελιξία σε επίπεδο κρατών μελών. Δηλαδή να δώσουμε τη διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη να επιλέξουν τον τρόπο που θα τον καταφέρουν. Στην Πολωνία η συμπαραγωγή ε, και θερμο, ο θερμοσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων είναι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε. Για τους τρεις στόχους που έχετε παρουσιάσει, το 20-20-20, μήπως θα ήταν καλύτερο να ορίσουμε τι ακριβώς σημαίνει αποδοτικότητα, γιατί δεν θέλουμε περιορισμούς. Θέλουμε πραγματική αποδοτικότητα, η οποία σημαίνει εξορθολογισμένη χρήση της ενέργειας. Μήπως θα έπρεπε να πεπλοκάρουμε και τις επενδύσεις, αυτές τις τεράστιες επενδύσεις που γίνονται σε μεγάλες μοναδές παραγωγής ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Νομίζω ότι η τεχνολογία CDS θα πρέπει να συγκρίνεται με άλλες τεχνολογίες σε άλλα καύσιμα γιατί θέλουμε να είμαστε δίκαια ανταγωνιστικοί. Ο κύριος Σίσλι. Η κυρία Σίσλι μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Η πρώτη μου ερώτηση σχετίζεται με τα όσα είπε ο συνάδελφος Οντί για τη συγκεκριμένη σχέση που υπάρχει μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ναμπούκο είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ο γογό South Stream, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια της ενεργειακής ευρωπαϊκής στρατηγικής. Για το South Stream μπορώ να σα πω πω η Ρωσία χρησιμοποιεί μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία είναι η εξή. Ε, θα τις επιτρέψει να μπει στην ε, ευρωπαϊκή αγορά απλώς με αυτά που προσφέρει. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε με ποιο, λόγο, ε, με ποιο τρόπο έχετε σκοπό να προστατεύσετε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και να καλύψετε τόσα έχουμε στο τρίτο πακέτο απελευθέρωσης. Η επόμενη ερώτηση είναι εξής. Αναφερθήκατε στη μακρά διαδικασία διοδότησης για τα ευρωπαϊκά έργα υποδομών, ενεργειακών υποδομών. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλάει για ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσει για τις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και θα ήθελα να μου πείτε και προσωπικά ποια είναι η γνώμη μας. Όπως επίσης με ενδιαφέρει η γνώμη σας για την αδειοδότηση των μονάδων παραγωγής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ευνοϊκό για τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν σκοπό να εισάγουν ε, την πυρηνική ενέργεια, αλλά και για τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν πολύ ε, μικρότερο δυναμικό, τουλάχιστον όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε και μια που είστε εδώ θα σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για τις διασυνδέσεις. Εσείς το είπατε, η διασύνδεση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε αυτή την, αυτό το στόχο μας που είναι η ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς, όπως επίσης και η διείσδυση της αγοράς, στην αγορά των, ε, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως το να γίνει αυτό ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεπεράσουμε τη συμφόρηση που έχουμε σε κάποια σημεία. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο να εφαρμόσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε ε, στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε τις πιο αδύναμες διασυνδέσεις που έχουμε στο ε, σύστημά μας. Και αναφέρομαι εδώ στις προσπάθειες που θα πρέπει να κάνουμε στο φυσικό αέριο. Γιατί εάν δεν συμφωνηθεί μεταξύ κρατών μελών, ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να παρέμβει Ε, ως διαμεσολαβητής στις επαφές αυτές και να παίξει ένα ρόλο παρόμοιο με αυτό που έπαιξε ο κύριος Μόντι στο παρελθόν ε, με την διασύνδεση της ηλεκτρικής ανέργειας. Πείτε μου λοιπόν, εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε σκοπό να παρέμβετε έτσι ώστε να αποσυμφορήσετε ε, αυτά τα σημεία συμφόρησης που έχουμε στο δίκτυό μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι καλύψαμε την ε, ομιλία, της ερωτήσεις, ε, αλλά ζήτησε η κυρία Τικάου ακόμη πολύ σύντομα να παρέμβει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα για τα μέτρα που σκοπεύει να πάρει η Κομισιόν για να καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλές οικογένειες, πολλά νοικοκυριά στην Ευρώπη, που είναι εκτεθειμένη, εκτεθειμένα στον κίνδυνο αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα μπορούσε να καλύψει το 4% της εθνικής ποσόστοσης. Αυτό το 4% μπορεί να δοθεί για να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων και κυρίως των κατοικιών. Των κατοικιών το τονίζω και το υπογραμμίζω αν θέλουμε να βελτιώσουμε την, την ενεργειακή τους ε, απόδοση. Και μην ξεχνάμε ότι το 99% των κτηρίων είναι χτισμένα στις αρχές του αιώνα, του προηγούμενου, και είναι ακόμα όρθια. Ε, πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με τον ε, συνάδελφό σας τον Επίτροπο, ούτω ώστε το 10% της εθνικής ποσόστοσης του ΦΕΝΤΕΡ να μπορέσει να δοθεί Δηλαδή το ποσοστό αυτό να δοθεί για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών, των σπιτιών. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ορισμένες ε, <clears throat> από τις ερωτήσεις ε, θα αντικατοπτριστούν και θα απαντηθούν στη συζήτηση που θα έχουμε για το road, μελλοντικό roadmap. Το, δηλαδή εστιάζουμε στη, στο μέλλον μέχρι το 2020 και η ασφάλεια, το μείγμα, το ενεργειακό, οι επενδύσεις έχουν πιο μακροπρόθεσμα ορίζοντα και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το συζητήσουμε όταν θα ξαναβρεθούμε του χρόνου το να γίνει συζήτηση άνετα χωρίς δία για να μπορέσουμε ε, να καλύψουμε όλο το θέμα. Όσον αφορά την ε, φτώχεια, ο Βέλγος ε, Υπουργός που προεδρεύει το Συμβούλιο, ο κύριος Μανιέτ, μας είπε ότι την Παρασκευή πρέπει να υποβάλουμε ένα έγγραφο το οποίο ε, θα καλύπτει ε, το κόστος ενεργείας, την φτώχεια ενεργείας και τι μπορεί να γίνει μέσω, με, με, ε, με μέσα πολιτικής αγοράς αλλά και διαφορετικά για να το επιλύσουμε διότι η ενεργειακή ε, ασφάλεια συμπληρώνει ή προκαλεί την διατροφική ασφάλεια και ε, γι' αυτό έχει σχέση με διάφορα στοιχεία και ε, επίσης ε, αν δούμε τις ε, επενδύσεις θα πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη συζήτηση του θέματος της ενεργειακής στόχιας. Όσον αφορά τους στόχους 2020-2020, αν μπορούμε να τους καταστήσουμε πιο ευέλικτους, καταρχήν πρέπει να τους αναλάβω και να τους εφαρμόσω διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν συμφωνηθεί πριν από την τρέχουσα περίοδο και όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακος και τις ανανεώσιμες ενέργειες είμαστε ακόμη στην αρχή των σκέψεών μας αλλά θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα λαμβάνοντας υπόψη τα κράτη-μέλη και χωρίς κάποιο δεσμευτικό χαρακτήρα, χωρίς κάποιον έλεγχο βασιζόμενοι μόνο εις την ευελιξία δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε διότι κάποια μέρα θα μας πούν τα κράτη-μέλη με συγχωρείτε δεν επιτύχαμε τους στόχους ε, ε, και το βλέπουμε από τους προϋπολογισμούς στα κράτη-μέλη αυτόν τον καιρό η πείρα μας είναι αρνητική η εμπιστοσύνη είναι καλή αλλά η εμπιστοσύνη και ο έλεγχος και ε, ίση στόχοι για όλους νομίζω ότι είναι ε, ο καλύτερος και ο πιο αξιόπιστος τρόπος ε, που υπάρχει για να προχωρήσουμε. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Ε, ε, η αποτελεσματικότητα σημαίνει εξοικονόμηση ή βελτίωση της ακριβίας της ενεργείας. Διότι πολλά αυτοκίνητα παραδείγματο χάρη είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από πλευράς ενεργείας τώρα από ό,τι πριν 20 χρόνια και χρειάζονται εξίσου πολύ βενζίνη. Διότι με καλύτερη αποδοτικότητα του κινητή μπόρεσε να απελευθερωθεί ενέργεια για το air condition του αυτοκινήτου, τον κλιματισμό δηλαδή, ε, για άλλα θέματα. Θέλουμε λοιπόν μία αύξηση της αποτελεσματικότητας ε, να υπάρξει στο 20% ή να εξοικονομηθεί κατά 20%. Είναι βασικό και πρέπει να το δούμε. Κύριε Τούρμες, τότε δεν πρέπει να μιλάμε για αποτελεσματικότητα διότι αυτό δεν το καταλαβαίνει κανείς και έτσι δεν πείθουμε τους πολίτες. Ε, όταν μιλάμε για εξοικονόμηση ενεργείας όλοι οι πολίτες παρακολουθούν ακόμη και τα παιδιά ξέρουν τι σημαίνει εξοικονόμηση. Αποτελεσματικότητα είναι μια ακαδημαϊκή ε, ε, σκοτεινή εικόνα την οποία κανείς δεν καταλαβαίνει. Όσον αφορά το χρόνο αναφορά σας συμφωνούμε και ε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, θα παραμείνουμε στο 2005 ή θα πάμε σε ένα νεότερο χρόνο αναφοράς. Επίσης οι προοπτικές, οι προοπτικές για τα ανεπτυγμένα κράτη-μέλη, για την, ε, ε, για την Ιταλία παραδείγματος χάρη μας δείχνει ότι χρειαζόμαστε ε, μία προοπτική όπου χρειάζεται περισσότερη ενέργεια και γι' αυτό στα πρότυπα τα οποία μου έχουν υποβληθεί και τα οποία δεν δέχομαι για τα κράτη-μέλη ακόμη και το Λουξεμβούργο που βρίσκονται στην ουρά για το χρόνο αναφοράς που χρειαστήκανε χωρίς αποτελεσματικότητα και χωρίς εξοικονόμηση ε, δεχόμαστε τα, την λογική ανάπτυξη αυξήσεως ε, της κατανάλωσης ενεργείας ε, χωρίς αυτά τα μέτρα εξοικονόμησης ή όχι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε μέχρι την Άνοιξη μαζί και αυτό έχει αναφερθεί και στην έκθεση του Κοινοβουλίου και γι' αυτό περιμένω την επόμενη εκθεσή σας διότι ξέρω ότι και εσείς ε, δεν συμφωνείτε ε, όλοι μεταξύ σας και οι συζητήσεις γίνονται επίσης ε, για τη διεύρεση λύσεων. Σχετικά με το South Stream, ο νοτικός διάδρομος Ναμπούκο Τάπ IGI είναι προς συμφέρον του Νότου και δεν θέλω εγώ να τον μπλοκάρω. Εγώ βλέπω ότι το South Stream είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τις κυβερνήσεις μας. Δηλαδή όταν έρχεται επίσκεψη από την ε, ε, Ρωσία στη Βιέννη, στην Σόφια, στο Βουκορέστι ε, απλώνουν το κόκκινο χαλί. Για το ευρύ θέμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οι ε, ε, χρηματοδότηση για το South Stream εκτός από την Gazprom είναι η SNDF, ε, η Ruhr Gas, Αυστριακή, ορισμένοι έχουν προσκληθεί και δέχθηκαν την πρόσκληση. Δηλαδή πρέπει να δούμε τις, τους συσχετικούς των δυνάμεων. Το ο, ο, Ναμπούκο είναι προς όφελος της Ευρώπης αλλά δεν θέλω να μπλοκάρω το South Stream. Και αν χρειάζεστε κάτι παραπάνω πέστε μου να το συζητήσω με τις κυβερνήσεις. Τους γνωρίζω όλους και θα δείτε ότι μπορούμε εδώ να καταρτήσουμε αρχές ακόμη και αν είναι αντίθετος ο άνεμος εκτός της αίθουσας μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα από ό,τι ίσως νομίζουμε. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε τα όρια μας και ε, μοιάζει με τον αθλητισμό. Εάν στο ύψος ε, ε, φάνεται στο 1,20 τότε μπορείτε να προπονηθείτε για το 1,40. Όχι όμως το 2,10 και ε, η υπερβολική φιλοδοξία μπορεί να είναι αρνητική αντί να είναι θετική η παρουσίαση η οποία προετάθη ε, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα κάνουμε εκθέσεις ε, για τις ε, βέλτιστες πρακτικές, για τα οικολογικά συστήματα, για συστήματα με πολλαπλά μέσα. Έχουμε κάθε εβδομάδα, νέ, κάθε εβδομάδα νέες προτάσεις και ε, απευθυνόμαστε στη δημόσια γνώμη. Αλλά δεν έχω ψευδεστήσεις. Πιστεύω ότι ο κύριος Φον Ρόμπο, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σαρκοζή, ο κύριος Γιούνκερ ε, δεν πρόκειται να εντυπωσιαστούν με τα καλοριφέρ που θα είναι στην ε, είσοδο. Λοιπόν, πιστέψτε με, εγώ δεν θέλω να γελιοποιηθούμε διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να συζητήσει σοβαρά θέματα. Πρέπει πέραν της, ε, ε, των ΡΟΜ της ε, Ελλάδος έχουμε ακόμη θέματα προς συζήτηση το, ως το Φεβρουάριο και αν δεν τα λύσουμε να ξεχάσουμε την ενέργεια. Εγώ όμως έχω αντιληφθεί τα προβλήματα και προς προσπαθώ να προωθήσω τις ε, νέες φάσεις της ενεργειακής πολιτικής τις οποίες θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις, πρέπει καταρχήν να υπάρχει εξυγίανση των κτηρίων και δεύτερον ανάπτυξη της υποδομής. Οπότε προγράμματα σαν τον Αμπούκο ή το Ίτερ όσο μεγάλα και να είναι θα αναπτυχθούν στο σωστό τους πλαίσιο. Εάν βλέπετε ότι σε κάθε μονάδα κατοικίας ε, η ε, ε, ενεργειακή εξυγίανση είναι μεταξύ 40 και 80.000 ε, ευρώ τότε αντιλαμβάνεσαι ότι το θέμα που μας απασχολεί η εξυγίαση των κτηρίων και η υποδομή θα αποτελέσουν τους πιο βασικούς, ε, τις πιο βασικές προκλήσεις χρηματοδοτήσεως για το μέλλον και δέχεται ε, έτσι να υπάρχει μία εξισωτική δικαιοσύνη διότι εάν τώρα επενδύσουμε στα ε, smart και στην ανανέωση των κτηρίων ε, και συγχρόνως θελήσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της ενεργείας και καλύτερη χρήση μέσα στον προϋπολογισμό και μικρότερο κόστος ενεργείας, τότε ε, θα μπορέσουν να υποφεληθούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας για τα επόμενα 30 έως 50 χρόνια. Άρα το θέμα της εξηγιάνσεως των κτηρίων και το θέμα της αποτελεσματικότητας και υποδομής είναι τα πιο βασικά θέματα για τα 20-30 επόμενα χρόνια κατά τρόπον ώστε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να έχουν κάτι αρκετά καλύτερο από ό,τι έχει η, η τωρινή γενιά και όσον αφορά τον προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα είναι οξύ θέμα έχουμε πάρα πολλά καλά προγράμματα ορισμένα λιγότερα λογικά και θα πρέπει να αξιολογηθούν και να διατυπώσουμε μία πρόταση για το πώς θα τα συνεχίσουμε τα Eurobonds είμαι ανοιχτός Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, εγώ ευχαρίστως να βρω χρήματα από όπου και να έρχονται, από τον προπολογισμό, από την τράπεζα, από τρίτους επενδυτές. Ε, θέλω να γίνει λογική χρήση. Ε, εάν πρόκειται για ίδιους πόρους ή ε, άλλους πόρους, αυτό δεν απασχολεί την ενεργειακή πολιτική, αλλά την δημοσιονομική και οικονομική πολιτική. Βλέπουμε εδώ το θέμα του προϋπολογισμού ε, για μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 και άκουσα και εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει πρόταση να προωθήσουμε τα Eurobonds οπότε ασχέτως της υποδομής ίσως δεν υπάρχει άλλος τομέας πλην της ενεργείας όπου μπορεί κανείς να αιτιολογήσει τη χρήση των Eurobonds και να το καταλάβει καταλάβουν και οι εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες μπορεί να πιστούν να ακολουθήσουν. Στη συνέχεια τέθηκε το θέμα του ΚΑΡΣ 21 εγώ πιστεύω ότι στο θέμα της ηλεκτρικής ε, ε, κινήσεως, το θέμα της μπαταρίας, το θέμα της πρίζας είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και θα είναι αποφασιστικά. Για τις πρίζες υπάρχουν οι λύσεις στις οποίες ορισμένοι ενδιαφερόμενοι έχουν ε, καθυστερήσει και ελπίζω ότι μέχρι την Άνοιξη θα διατυπωθούν προτάσεις αλλά από εκεί και πέρα ε, τα κράτη πρέπει να αποφασίσουν εάν θα δεχθούν τις προτάσεις της υπεύθυνη ομάδος. Στο θέμα των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας κύριε Τούρμες ε, δεν θέλω τίποτα να καταστρέψω. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την εξέλιξη των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια. Αλλά ο Γιος Καφίσερο, ο δικός σας κομματικός φίλος είχε προτείνει ε, το, την Ευρωπαϊκή ε, του δικαιώματος αποθηκεύσεως ε, της ανανεώσιμης ενέργειας και το πρόγραμμα προβλέπει μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει ε, με αυτόν τον τρόπο 15% του, της, του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρικού και πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για πενταροδεκάρες άρα πρέπει να δούμε ότι με το Μαρόκο, την Τινεσία, την Αλγερία και με άλλους υπάρχουν θέματα. Πρέπει να προωθήσουμε την, την υποδομή του Μαρόκου προς την την ε, ε, Ισπανία και από την Τινησία προς την Ιταλία κατά τρόπον ώστε να μην και με τα σκουπίδια πλέον στην Νάπολη όπως γίνεται και που δημιουργούν άλλα και πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε ηλεκτρικό με άλλους καλύτερους τρόπους. Το Ναμπούκο μπορεί ίσως να υπαρκέσει για μία αγορά. Εμείς σκεφτόμαστε και τους, τα μελλοντι, τους μελλοντικούς αγωγούς και άλλες συμφωνίες όσο ισχύει ακόμη το τρέχον πλαίσιο και γι' αυτό συμβουλευόμαστε όλα τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι ιδίως στον τομέα του αερίου το να είναι κανείς ανοιχτό στον ανταγωνισμό και το unbundling πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο και να το σεβαστούμε και στο μέλλον. Αυτά ήταν τα βασικά ερωτήματα που είχα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίσκοπε. Κύριε Τούρμες, ε, πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτηση γιατί έχουμε και άλλα θέματα, αλλά είναι δέκα δευτερόλεπτα, τρέχει το, ο χρόνος και σας ακούω. Χρειαζόμαστε λοιπόν, μια... έκθεση μισή ώρα όπου εμπειρογνώμονε από ένα εργαστήριο μπορούν να δείξουν ότι υπάρχει κάτι σε Σάντμπαϊ. Πρέπει να Πρέπει να σας πω πάντως ότι δεν κατάφερε ούτε να κλείσει τους διακόπτες και να τους βάλει στο stand-by για να το δούνε για να διακόψουν το κύκλο έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν το πείραμα. Οπότε επειδή ακριβώς είχε αυτό το πρόβλημα, τότε υποχρέωσε όλες τις κυβερνήσεις αυτός ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη μία αυτή δοκιμή να υιοθετήσουν τον κανόνα του ε, stand-by. Ε, Καταλαβαίνετε λοιπόν πως τέτοιου είδους επιδείξεις ή εκθέσεις ή δοκιμές ε, πείθουν τους πολιτικούς. Ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε καλή εμπειρία και ίσως μπορεί όπως και ο κύριος Μπούς που τότε επίστη να πιστούν και οι δικοί μας πολιτικοί. Ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στον ε, Επίτροπο να απαντήσει. Ε, χαίρομαι αν ε, έγινε αυτό με τον κύριο Μπούς, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι θα συζητήσω με τον Ούγγρο Υπουργό Ενεργείας εάν δεν θα μπορέσουμε στο θέ... στη συζήτηση για το Συμβούλιο Ενεργείας της Ανοίξεως να κάνουμε μία μικρή έκθεση σχετικά με την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Βέβαια εγώ δεν είμαι ο, υπο, είναι η Ουγγαρία, είναι ο κύριος Φων αλλά μπορώ να προσπαθήσω σε λίγο χρόνο να το επιτύχω. Θα το σημειώσω και ίσως μπορέσουμε να κάνουμε ε, μία μικρή έκθεση για την αποτελεσματικότητα ενέργειας ε, μέσα στο ιδιωτικό σπίτι, στον νοικοκυριό για την ψήξη και τη θέρμανση. Σας ευχαριστώ και ε, προσβλέπω στην έκθεση. Θα ήθελα όμως καταρχήν ε, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο εν ονόματί σας, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Όσοι ε, αυτή τη στιγμή μιλούν παρακαλώ να χαμηλώσουν τους τόνους. Ε, τον... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η ώρα είναι προχωρημένη. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ λακωνικός και γρήγορος. Πρόκειται για τη διαδικασία αναθεώρησης της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μέγιστα επιτρεπά, επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές μετά από πυρηνικό ατύχημα ή μετά από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Συνήθως αυτό γίνεται στα πλαίσια μιας διαδικασίας διαβούλευσης. Ε, παραπέμπουμε στα άρθρα της συνθήκης ε, Euratom. Ε, στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων που κάναμε στην Επιτροπή μας, επειδή υπήρχε αυτό το θέμα με τα άρθρα της Euratom, μιλήσαμε για την νομική βάση. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να θίξουμε σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη νομική βάση, όχι το άρθρο 31 Euratom, αλλά να βασιστούμε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Να διαλέξουμε δηλαδή ένα άρθρο από τη συνθήκη της Λισαβόνας ως νομική βάση. Καταρχάς, εν Φυσικά ήρθαμε σε επαφή με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και χάρη στην ε, πρωτοβουλία σας, κύριε Πρόεδρε, ε, ήρθαμε και σε επαφή με τον ε, πρόεδρο Λένε της ε, αρμόδιας επιτροπής, της νομικής επιτροπής και ομόφωνα ε, συμφωνήσαμε να περάσουμε από τη συνθήκη Euratom στην συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε από τη διαβούλευση στην συναπόφαση, δηλαδή δύο διαφορετικές διαδικασίες και το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό, πολύ διαφορετικό. Αυτή είναι και η θέση του Κοινοβουλίου. Ε, θέλουμε να, το, να την προτάξουμε αυτή η θέση στην έκθεση αυτή και βασιζόμαστε στη συνένεση όλων των μελών της Επιτροπής μας. Ε, φυσικά η θέση του Συμβουλίου είναι διαφορετική, λογικό είναι. Και η Κομισιόν έχει και αυτή την ε, δική της άποψη για το θέμα αυτό. Αυτό τι σημαίνει, Πρόεδρε. Χωρί να μπω τώρα σε λεπτομέρειε για όλε τι ε, τροπολογίε που είναι καμιά εβδομηνταριά, δεν μπορώ να τι διατρέξω όλε, αλλά μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσει και βεβαίω και η Κομισιόν είναι εδώ για να απαντήσει σε σχετικέ ερωτήσεις. Θέλω μόνο να μιλήσω για τα πιο σημαντικά άρθρα, το άρθρο 2, Φερρυπίν, το οποίο το έχουμε προσαρμόσει από την αρχή μέχρι το τέλος με την βοήθεια των συναδέλφων και προτείνουμε η Κομισιόν σε περίπτωση που υπάρξει ατύχημα να πάρει από την αρχή την απόφαση να καθορίσει τους ε, κατάλληλους κανόνες και να τους θέσει σε εφαρμογή πάρα αυτά, αμιλητή. Γιατί ξεκινάμε από την υπόθεση ότι πρόκειται για αρμοδιότητες εκτελεστικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε τις αρμοδιότητες αυτές, να τις δώσουμε στην Επιτροπή και δεν θα πρέπει να περάσουν στο Συμβούλιο. Ε, ένα άλλο σημείο που συνδέεται με το προηγούμενο και το συμπληρώνει, προτείναμε μια νέα τροπολογία στην, ε, στο άρθρο 5. Ε, το αναφέρω. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα, αυτή στιγμή που υπάρξουν νέα δεδομένα, νέες γνώσεις, προτείνουμε μέσω της ε, εξουσιοδότησης να εκχωρήσουμε αυτές τις αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτής της πράξης κατά εξουσιοδότηση να αποφασίσει για την εφαρμογή αυτών των νέων δεδομένων. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ένα τμήμα των αρμοδιοτήτων περνάει εκ νέου από το Συμβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι ανεφόρων φυσικά. Φυσικά απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μια έκθεση, να την παρουσιάσει και στο Κοινοβούλιο και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου ε, είναι ότι μπορεί να εκ νέου να ξαναπάρει πίσω αυτές τις αρμοδιότητες, να τις φετεριστεί αν θέλετε, να τις πάρει πίσω. Επίσης, κυρώσεις σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν σέβεται τον ορισμό για τα τρόφιμα, για τα πολύ μικρά παιδιά, για τα μωρά μάλλον. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί όπως σας είπα στέκομαι στα πιο βασικά στοιχεία της έκθεσης. Ε, τα πιο βασικά στοιχεία είναι στις, στο παράρτημα. Κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο παράρτημα 1, το βασικό παράτημα για τα βασικά τρόφιμα, και τα τρόφιμα προτεραιότητας, τα, το παράρτημα 2, τα λιγότερο σημαντικά τρόφιμα και το τρίτο ε, παράτημα που αφορά τις ζωοτροφές. Τώρα, οι τροπολογίες ε, από τους συναδέλφους είναι ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν οι τιμές της ραδιενέργειας και παραπέμπουμε στο μοντέλο της οργάνωσης FDA, της Αμερικάνικης ε, αυτής υπηρεσίας, όπου οι συνάδελφοι λένε ότι οι κανόνες αυτή της FDA είναι πολύ πιο αυστηροί από τους δικούς μας. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις βέβαια για το θέμα αυτό και προτείνω να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το θέμα, γιατί αυτό είναι εμπειρογνώμονας για αυτά τα θέματα. Μπορούμε να ακούσουμε τη γνώμη του λοιπόν. Υπάρχουν ε, και άλλες προτάσεις υπομορφή ε, τροπολογιών που προτείνουν ρητάν το παράρτημα για τα λιγότερο σημαντικά τρόφιμα να διαγραφεί και όλα τα τρόφιμα που υπάρχουν στα διάφορα παρατήματα να τοποθετηθούν στο παράρτημα 1. Να θεωρήσουμε δηλαδή ότι όλα τα τρόφιμα είναι προτεραιότητας και να... ότι πρέπει δηλαδή να ανταποκρίνονται σε πιο αυστηρές προδιαγραφές. Επίσης, έχουμε αυτές τις τροπολογίες που ουσιαστικά προτείνουν την μεταφορά των τροφίμων από το πάρτιμα 2 στο πάρτιμα 1. Όπως σας είπα, υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία δεν, ε, έχουμε, δεν τα έχουμε ρυθμίσει. Έχουμε ακόμα μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Θέλω να ακούσω την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έχουμε, όπως σας είπα, ε, την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να βρούμε και συμβιβαστικές ε, τροπολογίες ή συμβιβασμούς. Ο Κλοντ Τούρμες. Ο Μισελ Ριβάζη είναι ο σκιώδης μας εισηγητής ή σκιώδης εισηγητριά μας. Παρουσιάζω τη θέση της Ευχαριστώ, κύριε Μπελέτ, για την παρουσίασή σας. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, πρότεινε τη μεταφορά στην άλλη νομική βάση, να χρησιμοποιήσουμε την άλλη νομική βάση. Καλό είναι αυτό. Το άλλο θέμα που αναφέρατε είναι να αναλύσουμε τους κανόνες που παρουσιάζονται και οι οποίοι δεν έχουν ε, εξυγχρονιστεί από το 89. Έκτοτε όμως έχουμε νέα επιστημονικά στοιχεία για τη σχέση μεταξύ της ραδιενέργειας και της υγείας. Ε, Παραδείγματο χάρη, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν, ας πούμε, ε, σε, κοντά σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, ε, αυτοί απολάβουν αυτών των νέων κανόνων, ενώ η δική μας νομοθεσία υστερεί ε, σε σχέση με τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε. Επίσης το άλλο που αναφέρατε για τις ΗΠΑ Πολιτείες και για την παγκόσμια, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έχουν άλλους κανόνες. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον πιο ευπαθή πληθυσμό, λένε αυτοί. Ε, στις δικές μας προτάσεις προτείνει η Κομισιόν γίνεται ε, διάκριση ανάμεσα στα παιδιά και στους ενήλικες. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η διάκριση, να πάρει οργή. Αν πας στο σούπερ μάρκετ δηλαδή και αγοράσεις φαγητά, θα πρέπει να δώσεις στα παιδιά σου κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που τρως εσύ. Αυτό δεν γίνεται, δεν είναι πρακτικό. Γι' αυτό νομίζω ότι πιστεύω πως πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τη δική μας νομοθεσία με τα διεθνή πρότυπα και να υιοθετήσουμε, να ενστερνιστούμε την προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την επόμενη συνεδρία των σκιωδών εισηγητών, ούτω ώστε να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Ναι. Oui, euh, donc euh, plusieurs Ακούστηκαν πολλές ε, ερωτήσεις. Μου ζητήσατε λοιπόν να λάβω το λόγο, θα το κάνω, κάνοντας κάποια γενικά σχόλια. Λαμβάνοντας βέβαια και υπόψη τα είπε ο κύριος Τουρμές και ο κύριος Μελωτό εισηγητής. Ήταν σχόλια για τις τροπολογίες και θα τα απαντήσω όλα μαζί. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω όλες τις τροπολογίες που είναι σχετικές με τη νομική βάση και τα νομική σχέση θέματα. Δεν υπάρχει λόγος να μιλήσετε για τις τροπολογίες. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε και αργότερα. Λοιπόν, για την νομική βάση φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βέβαια θα δούμε τις εξελίξεις έχουν τελείως διαφορετικές θέσεις για το σημείο αυτό. Να σας υπενθυμίσω όμως το κείμενο του 106α εδάφιο 3 της Ενοποιημένης Συμφωνίας ε, Euratom είναι το παλιό 305 για τους κανόνες Euratom και πώς αυτοί μπορούν να συμμορφωθούν με τους κανόνες που έχουμε στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους εφαρμοστικούς κανόνες λειτουργίας. γιατί εκεί δεν έχουμε καμία παρέκκληση από τις διατάξεις της συνθήκης Ευρατών. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό που πολύ συχνά έχουμε πει στο παρελθόν είναι από τη στιγμή που η συνθήκη Ευρατόμ είχε τις απαραίτητες αρμοδιότητες για να εγκρίνει μέτρα, η συνθήκη αυτή, η εξειδικευμένη αυτή συνθήκη εφαρμόζονταν και θα εφαρμόζεται ως ο ειδικό νόμος. Για την νομική βάση λοιπόν δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Για τις τροπολογίες. Εδώ έχουμε κάποια πιο τεχνικά θέματα. Αρκετές τροπολογίες, όπως μας είπε ο κύριος Τουρμές, λένε πως η αξία αυτού του κανονισμού θα με συγχωρείτε πως ο κανονισμός θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί, να έχει εξυγχρονιστεί και αυτό δεν έχει συμβεί από τη στιγμή που εγκρίθηκε. Από το 1995 λοιπά που είχαμε την έγκριση της νομικής βάσης, που ήταν η οδηγία που όρισε τους βασικούς κανόνες, την 86-29 ευρατών από την οδηγία αυτή λοιπόν και μετά, η μείωση της ετήσιας δόσης από τα 5 στα 1 λυσιβέρ. Και αυτό για το ευρύτερο κοινό. Από τότε λοιπόν η ομάδα εμπειρογνωμών κάθε χρόνο εξετάζει τα αποδεκτά ανώτατα όρια που ορίζονται μέσα στον κανονισμό. Άρα λοιπόν ουσιαστικά πρόκειται για νέα όρια, για νέα ανώτατα όρια, μια που είναι αυτές οι δόσεις, αυτοί οι περιορισμοί στην ανώτατη δόση, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό το ανώτατο επιτρεπτό ε, όριο για την ε, ε ακτινοβόληση, για τα τρόφιμα. Αυτό γιατί το κάναμε, γιατί θέλαμε ένα περιθώριο ασφαλείας και πρέπει να σας πω από το 1987 έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι εμπειρογνώμονες ε, συμβούλευσαν την, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς βάλαμε βασιζόμενοι στα λεγόμενά τους μια πρόταση και η πρόταση αυτή ήταν πάρα πολύ αυστηρή, δηλαδή είχε εντάξει διάφορα όρια ασφαλείας και για κάποια ραδιονουκλεΐδια τα ανώτατα όρια τα διέρεσε για το 3 ή για το 4 για να είναι ακόμα πιο σίγουρο. Έτσι λοιπόν το 1995 κοιτάξαμε αυτά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και είδαμε αν αντιστοιχούν πάντα στους κανόνες είτε της Ευρατόμ είτε στους διεθνείς κανόνες, γιατί οι κανόνες Ευρατόμ ουσιαστικά ε, ακολουθούν τις ε, διεθνείς οδηγίες ε, που δίδονται από την Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη Ραδιενέργεια. Το 2006, και αυτό είναι κάτι το επιπρόσθετο. Παρόλο που είχαμε ξεκινήσει εργασία στο 4 ή το 5, η Επιτροπή Κότεξ Αλιμεντάριος, που δεν που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, έθεσε νέα όρια ε, για τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στο διεθνές εμπόριο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εντολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την αρχή μέχρι το τέλος συμμετείχε σε όλες τις εργασίες που κάνει αυτή η Επιτροπή η οποία ανήκει κυρίως στον ΦΑΟ και χρησιμοποίησε τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποίησε για να προετοιμάσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες για να κάνει τους υπολογισμούς της και για να ορίσει αυτά τα ανώτατα όρια που επαναλαμβάνω όπως είπατε και εσείς δεν είναι τα ε, είναι δεσμευτικά γιατί είναι κατευθυντήριες γραμμές για τον ορισμό αυτών. Τώρα το ότι υπάρχουν διαφορές, ναι. Στην Επιτροπή Κόντεξ Αλιμεντάριους δεν θέλανε να πούνε 2.500 ή 400 μπεκερέλ ένα κιλό. Θέλανε να έχουν ε, ένα σύστημα που θα λέει 1, 10, 100. Κοιτάξτε, είχαν τα τρόφιμα για βρέφη και είχαν και τα γενικά τρόφιμα, αλλά δεν είχαν όλες τις κατηγορίες που έχουμε εμείς. Επίσης, τα ραδιονουκλίδια τα κατηγοριοποίησαν με τον τρόπο που κάνουμε εμείς. Εμείς ε, ε, για τα στοιχεία αυτά λαμβάνουμε υπόψη το θέμα της ευαισθησία τους. Αλλά βέβαια καταλαβαίνετε πως πολλές φορές κάποιο γλιστράει, ξεγλιστράει σε κάποια άλλη κατηγορία. Αυτό συμβαίνει. Ε, επαναλαμβάνω όμως πως οι υπολογισμοί μας βασίστηκαν στα ίδια στοιχεία Και βέβαια έχουμε τα διάφορα ποσοστά των τροφίμων, για παράδειγμα, που καταναλώνται και είναι κοντά στα όρια και κάποιες άλλες τέτοια περιπτώσεις, αλλά νομίζω πως εμείς και αυτοί χρησιμοποίησαν τα ίδια όρια, τα οποία επαληθεύτηκαν το 1995, που ήταν το 1 μιλισιβέρ. Ήθελα να σας υπενθυμίσω γιατί μέσα στις τροπολογίες εσείς αναφέρεστε σε πολλές επιτροπές και παντού διαγράφεται την ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχουμε στο άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ. Και πρέπει να σας πω πως αναφέρεται κάπου και στα στοιχεία αυτής της ομάδας δεν είναι επαρκώς διάφανα. Η Επιστημονική Επιτροπή που επικαιρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μόνη η οποία έχει την επαρκή ε, πραγματογνωμοσύνη ε, για τα θέματα της ε, ραδιενέργειας. Και αυτή η πραγματογνωμοσύνη δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να βρεθεί και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων. Όποτε έχουν πρόβλημα με ε, όρια ραδιενέργειας, είτε έρχονται σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, είτε με το τμήμα μας απευθείας και μας θέτουν το ερώτημα, για παράδειγμα, τι επίπεδο ευαισθησίας έχουμε, για παράδειγμα, όπως είχαμε με το ουράνιο στο πόσιμο είδωρ, είτε με την ε, ε, χημική τοξικότητα κάποιων στοιχείων ή τροφίμων, μας στέλνουν αυτά τα ερωτήματα, τα οποία εμείς απευθύνουμε μετά στην Επιτροπή Άρθρου 31, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι η, η, η αυθεντία στο χώρο αυτό. Και μάλιστα ε, αποφασίζει την παράταση ή όχι του κανονισμού που δεν απορρέει από τη συνθήκη ε, Ευρατόμ. Όταν μιλάμε για τις εισαγωγές, από παράδειγμα, συμφωνίες που ε, διέπονται από ε, άλλους κανονισμούς. Λέτε, εισαγωγές προϊόντων, κομιτολογία, παράταση ή όχι του καθεστώτος. Στην περίπτωση τι και πάλι συμβουλευόμαστε την Επιτροπή άρθρου 31 και για το κατά πόσο είναι διάφανες οι εργασίες της, θα ήθελα να προσθέσω εδώ πως τα ονόματα και οι ιδιότητες των μελών αυτής της Επιτροπής είναι στη διάθεσή σας, βρίσκονται στο site μας στο ίντερνετ ε, και μπορείτε να τα δείτε από εκεί. Και έχει επίσης ένα εσωτερικό κανονισμό που έχει και κάποιους δεοντολογικούς ε, κανόνες για να εξασφαλίσουν τη λειτουργία της. Σε πολλές τροπολογίες λοιπόν αναφέρεται πως τα ανώτατα επιτρεπτά όρια θα πρέπει να βασίζονται στις απαιτήσει προστασίας πληθυσμών ε, που βρίσκονται στην πιο κρίσιμη και στην πιο, των πιο τροτών πληθυσμών, ε, αυτών που βρίσκονται στην πιο κρίσιμη κατάσταση. Τι, μιλά, τι σημαίνει σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν είναι λογικό να ρυθμίζει κανείς την αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τρόφιμα βασιζόμενοι στην ομάδα που έχει τα πιο κρίσιμα προβλήματα, η οποία ενδεχομένως έχει αυτάρκεια σε ε, τρόφιμα, για παράδειγμα αυτοκατανάλωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον γενικό πληθυσμό, όχι κάποιες ε, περιορισμένες ομάδες. Παρόλα αυτά η Κομισιόν έχει εκδώσει συστάσεις συστάσεις βασιζόμενοι στην, στο άρθρο 38 της Συνθήκης Ευρατών που δίνει αυτή τη δυνατότητα και μετά το ατύχημα στο Τσερνόβιλ για τα άτομα τα οποία καταναλώνουν πολλά προϊόντα δασικά, δηλαδή άγρια μανιτάρια, άγρια μούρα, ε, κυνήγι. Άρα λοιπόν λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες αυτών των ατόμων. Αυτό για τους, τους κρίσιμους πληθυσμούς. Τώρα, για τους πιο ευάλωτους ή τροτούς πληθυσμούς, εδώ έχω να σας πω το εξής. Η κατάρτιση ανώτατων τιμών που, έχουν, που έχει κάνει η Επιτροπή άρθρο 31 και η οποία προχώρησε σε υπολογισμούς για διάφορες ηλικιακέ ομάδες. Είδα όλα λοιπόν τα ραδιονουκλίδια, είδα όλα τα καθεστώτα και έκανε κάποιους υπολογισμούς έλαβε υπόψη τις καταναλώσεις και πήρε τρεις ηλικιακέ ομάδες. Ενό έτου, δέκα ετών και ενήλικέ. Και σε κάθε μία περίπτωση, στο εσωτερικό αυτής της ομάδας της ηλικιακή διατήρησε τι πιο αυστη... τις πιο αυστηρές τιμές, τις πιο χαμηλές δηλαδή, και αυτές είναι οι ανώτατες τιμές ή τα όρια τα οποία εμφανίζονται στον κανονισμό. Και θα προσθέσω εδώ πω όντω έχουμε συγκεκριμένες τιμές για τα τρόφιμα για τα βρέφη, για τα νήπια. Εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε. Ναι. Υπάρχει ειδική τροφή. Εσείς μιλήσατε για παιδιά, για τα βρέφη. Εγώ μιλάω για βρέφη, για νήπια. Και αυτή τη στιγμή στο εμπόριο κυκλοφορούν τρόφιμα που απευθύνονται στα βρέφη. Τώρα, τι σημαίνει τρόφιμα για βρέφη μέχρι τους 4 μήνες, μέχρι τους 6 μήνες, μέχρι τους 12 μήνες. Νομίζω ότι αυτό εντάξει θα μπορούσαμε να το δούμε. Έχουμε λοιπόν το πιο αυστηρό, την πιο αυστηρή τιμή για κάθε ηλικιακή ομάδα και αυτήν την τιμή την εφαρμόσαμε σε κάθε περίπτωση εκτός από τα νήπια ή βρέφη. Γιατί για τα ενός τι να σας πω, ε, νομίζω ότι προστατεύουμε και τους ενήλικες με τον ίδιο τρόπο που προστατεύουμε και αυτές τις πολύ μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Και μπορεί με αυτή η προσέγγιση να μην έχει συμφωνηθεί από όλους, αλλά τουλάχιστον ακολουθεί μια συγκεκριμένη λογική. Κάποιες τροπολογίες δίνουν την εντύπωση πως θα πρέπει να τηρήσουμε πιο ενήμερο τον πληθυσμό, το κοινό και πως μακροπρόθεσμα και νομίζω είναι η κυρία Ριβάζη που υπέβαλε αυτές τις τροπολογίες, θα πρέπει να συμμορφωθούν με το επίπεδο έκθεσης της οδηγίας 9629 ε, της Ευρωματό στο θέμα αυτό. Να σας πω το εξή. Θα πρέπει βέβαια να τηρήσουμε ενήμερο το κοινό. Όμως υπάρχει σχετική οδηγία η 618 του 86 της Ευρατόμ για τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που εφαρμόζονται πριν από κάποιο ατύχημα ή κάποιο έκτακτο περιστατικό, όπως επίσης και ε, το τι, πώς θα πρέπει να δράσουμε σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού έκθεσης ραδιενέργεια. Συνδέεται επίσης με αυτό που λέγεται αργότερα, πως θα πρέπει η αναφορά, ε, η παραπομπή στην οδηγία ε, που θέτει τα, τις βασικές αξίες θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρη. Εγώ θα πω το αντίθετο, όχι μόνο μακροπρόθεσμα, αλλά συνέχεια. Γιατί οι τιμές που έχουμε στον κανονισμό και τις οποίες εσείς εξετάζετε και αναθεωρείτε, απορρέουν από την οδηγία. Και το είπα προηγουμένως. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τις υπενθυμίζουμε συνέχεια στον κανονισμό μας. Και τέλος, θα κλείσω λέγοντας πως η προστασία από τη ραδιενέργεια βρίσκεται λοιπόν στα άρθρα 39 και 38 στο κεφάλαιο 3 της συνθήκης Ευρωτόμ, Και βεβαίως μην ξεχνάτε και το άρθρο 2β. Είναι ένα πρωταρχικό δικαίωμα το οποίο ε, συνδέεται με ένα παράγωγο δικαίωμα και θα σας δείξω εδώ το κείμενο που βρίσκεται σε, μια, σε ένα τόμο 250 σελίδων. Ίσως αυτό μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω με ε, ε, ιδιωτικές ε, συζητήσεις διότι θα έπρεπε να τελειώσουμε τώρα ο κύριος Τούρμες έχει ακόμη μία ερώτηση και οι διερμηνείς θα φύγουν λέει ο πρόεδρος Πρωτογενές δίκαιο ε, δευτερογενές ο κανονισμός με τα ανώτατα όρια σε περίπτωση ατυχήματος όλα αυτά τα βρίσκεται σε αυτό το κείμενο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λόντ Τούρμες, θέλω να απαντήσω σε αυτή την παρουσίαση τύπου Βολτέρου που συχνά ε, χρησιμοποιούν αυτοί που δουλεύουν με, τα, μετρα και με αυτά τα θέματα. Εγώ έχω τον κανόνα πόσα μπεκερέλ ανά είναι 10 ανά 100 χιλιάδες. Και στα παρατήρηματά σας έχετε τα σχετικά νούμερα. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες για κάποια από αυτά που είπατε. Σήμερα δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Προτείνω να οργανώσουμε μία πιο τεχνική συνεδρίαση για να αντιπαρατεθούμε. Να δω πώς θα απαντήσετε στις αμφιβολίες που έχω ε, και να δω τι πληροφορίες θα μας δώσει η Κομισιόν. Γιατί εγώ αμφιβάλλω για αυτές τις πληροφορίες που μας δίνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε μία τεχνική συνεδρίαση. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ξανασυνεδριάσουμε επί του θέματος και να προετοιμαστούμε για την ψηφοφορία και ο κύριος Μπέλε πολύ καλά προχώρησε ε, ε, διευκρινίσαμε τα βασικά θέματα, τα υπόλοιπα θα συζητηθούν ε, κατά την ψηφοφορία αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ και τα υπόλοιπα αύριο το πρωί.